Wznawiam posiedzenie. Protokół z wczorajszego posiedzenia. Συνεχίζεται τη Τα χθεσινά πρακτικά έχουν ε, διανεμηθεί. Υπάρχουν σχόλια, φαίνεται πως όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι τα χθεσινά πρακτικά έχουν εγκριθεί.